Pan Przewodniczący! Colleagues, please take a seat. Please take a seat. Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θλιβερά μαντάτα έχω για σας. Let me say few words, colleagues. Να πω δύο λόγια σχετικά, συνάδελφοι. This is sad information. Mr. Angelo Vassallo. Ο κύριος Άντζελο Βασάλο, 57 ετών, δήμαχος στην περιοχή Καμπάνια στην Ιταλία, δολοφονήθηκε την Κυριακή το βράδυ από την Καμόρα, καθώς βρισκόταν καθοδόν να επιστρέψει σπίτι του ήταν καλύτερα γνωστός ως ο περιβαλλοντικός ε, δήμαρχος για τις προσπάθειές του να βοηθήσει για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στην περιοχή του. Πάντα αγωνιζόταν κατά της διείσδυσης ε, του οργανωμένου εγκλήματος στην πόλη του. Είχε πραγματικά πολύ μεγάλη ανθρωπιά και πολύ μεγάλη επαφή με τους πολίτες του. Δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε τον ρόλο του οργανωμένου εγκλήματος σε κάποια από τα κράτη-μέλη μας θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι αλληλέγγυοι ώστε να μπορέσουμε να ξεριζώσουμε αυτή τη μάστιγα από τις κοινωνίες μας ώστε ο, ο θάνατος του Άντζελο Βασάλο να μην έχει πάει ε, του κάκου. Θα ήθελα να ε, εγερθούμε και να αποτίσουμε ενός λεπτού φωτιμή σας στη μνήμη του. Παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Τώρα αγαπητοί συνάδελφοι προχωρούμε στις ψηφοφορίες που έχουμε. Ο κύριος Καρίν βλέπω έχει διαδικαστικό παρακαλώ. Mr. President, thank you. 48... Πρόεδρε ευχαριστώ. 48 ώρες ε, από σήμερα θα ε, έχουν ε, τη γιορτή τους ε, του ε, ΕΒ μετά το τέλος του Ραμαντάν και έχει προγραμματιστεί να το κάψιμο του Κοράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πράξη έχει καταγγελθεί και από την κυβέρνηση, τον είπα και από το Βατικανό. Ελπίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα καταδικάσει αυτό το εγχείρημα εξίσου. είναι η πράξη, η δράση ενός ατόμου και των οπαδών του το κάψιμο του Κορανίου και δεν πρέπει η πράξη, η πράξη αυτή να ταυτιστεί με τη Δύση ή με τη Χριστιανοσύνη και να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα αυτός ο πάστορας με το κάψιμο του Κορανίου. Έχει απομονωθεί ήδη. Μόνο μέσω οποιασδήποτε ε, αντίδρασης ε, μπορεί κάποια τέτοια ε,